που διεκόπη στις 12 Μαρτίου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναλαμβάνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όλοι είμαστε βεβαίως συντετριμένοι